Vamos a empezar la, la sesión. Ας αρχίσουμε. Καλησπέρα σας σε όλες και όλους. Πρώτον, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, αλλά προηγουμένως έγκριση των πρακτικών. 4 και 5 Μαΐου 2015. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνονται τα πρακτικά. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι σίγουρα το σημείο 5 και 6 θα καθυστερήσει ε, μάλλον θα αναβληθεί διότι δεν συμφώνησε το Προεδρείο και ό,τι έχει να κάνει με το Τουρκμενιστάν αναβάλλεται. Θα το ξαναπώ στη συνέχεια αυτό. Λοιπόν, α αρχίσουμε όμω με την ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή του προπολογισμού Χωσέ Μανουέλ Φερνάντε, που είναι ο εισηγητής για το προπολογισμό του 2016. στι 27 Μαου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το προσχέδιο ε, του προπολογισμού και σίγουρα εργάζεται εντατικά ο κύριος Φερνάντες. Η συζήτηση αυτή που έχουμε τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να κάνει η Επιτροπή μας τη φωνή της να ακουστεί και να ζητήσουμε επαρκή κονδύλια για τις ε, εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο. Αλλά βασικά σήμερα θέλουμε να συλλέξουμε εντυπώσει να βολιδοσκοπήσουμε προς τα που πηγαίνουν οι συζητήσεις για την εκτέλεση αυτή. Έχει απόλυτη σημασία και είναι ουσιαστική ε, ε, η χρηματοδότηση, ε, η επαρκής χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων για να έχουμε τη δυνατότητα ανεξάρτητα να δραστηριοποιούμε θανά τον κόσμο. παρακαλώ λοιπόν κύριε Φερνάντες, εξηγήστε μας. euh, στη σύνθεση. Ε, ε, ακούτε, συγγνώμη. Ήθελα μόνο να ζητήσω για το Τουρκμενιστάν. Τι θα γίνει. Εγώ είμαι σκιώδης ηγητής. Δεν ξέρω, έχετε καμιά εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. Αναβάλλετε για πότε δηλαδή και τι συμβαίνει. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα. Και για ποιο λόγο ελήφθη αυτή η απόφαση. Θέλετε να μα πείτε. Bueno, yo, eh, la información que tenemos es que no se Κοιτάξτε, έχουμε την εξή προφόρηση ότι στο Προεδρείο, στη συνεδρία των συντονιστών δεν συζητήθηκε. Θα συζητηθεί την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε ακριβώ για πότε αναβάλλεται. Πάντω αυτό που ξέρω είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το αναβάλουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Perdone, disculpe. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήρθα να παρουσιάσω τις κύριες κατευθυντήρια γραμμές μας. Γιατί την περασμένη εβδομάδα, 20 με 27, έκανε την πρόταση της σχεδίου προϋπολογισμού η Κομισιόν. Γενικά σας υπενθυμίζω ότι ο στόχος μας είναι τα τρία, ή τρεις στόχοι επιχειρήσεις, απασχόληση κλπ. Και το επιχειρησιακό ή επιχειρηματικό πνεύμα. Αλλά βάλαμε και τέταρτο την εσωτερική και εξωτερική αλληλεγγύη. Άρα στο τμήμα 4 βάζουμε στις κατευθυντήριες γραμμές μας και αυτή την προτεραιότητα. Επίσης κάτι άλλο που βάλαμε στο ψήφισμα που δεν θα έπρεπε να το είχαμε βάλει γιατί είναι αυτονόητο. Υπενθυμίζουμε προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο ότι πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι συμβιβασμοί και οι δεσμεύσει των μεν και των δε όπως τον πολιετή χαρακτήρα του πολιτισμού κλπ. Δηλαδή οι συμβιβαστικές προτάσεις, οι συμβιβασμοί πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Επίσης όμως πρέπει να χορηγηθούν τα κονδύλια για τις προβλέψεις και την χρήση των αποθεμάτων ή που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Ε, στο καινούργιο άρθρο 14 λέμε τα κονδύλια, τα, οι προβλέψεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιο χρόνο να μπορούν μετά να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη, για την απασχόληση να τα, επαναλάβ, τα επαναλαμβάνουμε αυτά γιατί το Συμβούλιο δεν θέλει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρησιμοποιητά κονδύλια και άρα στην ουσία θέλει να μειωθεί ο προϋπολογισμός να έχει περικοπάσα. Αλλά το Κοινοβούλιο επειδή επιμένει στην ευελιξία ευελιξία επιμένει να χρησιμοποιηθούν και τα χρησιμοποιητά κανδύλια. Όπως ξέρετε σε λίγο θα υποβληθούν τα νέα πιλωτικά προγράμματα 4 Ιουνίου μάλιστα. Στις 17 Ιουνίου λίγη προθεσμία για την έγκριση των εντολών για τον τριμερή διάλογο. Μέσα Σεπτεμβρίου από κανένα λογισμό για τον Οκτώβριο, 27 και 29 Σεπτεμβρίου και 30. Ψήφισμα για τις τροπολο... ψήφιση των ε, τροπολογιών για τον προπολογισμό, μετά τον Οκτώβριο Ολομέλεια, ε, Οκτωβρίου, Νοέμβριο η συνδιαλλαγή και αυτά ήταν το χρονοδιάγραμμα αν καταλάβατε. Η πρόταση της Κομισιόν Τώρα μιλάω για το, για το σχέδιο του, της 27ης της Κομισιόν, της περασμένης εβδομάδας δηλαδή. Είναι καλό σχετικό σχέδιο, θετικό και για το τμήμα 4. Βλέπουμε δηλαδή ότι τους ενδιαφέρει να γίνουν σεβαστοί οι συμβιβασμοί όπως έλεγα και πριν. Και χάρη σε αυτό υπάρχει μια σημαντική αύξηση των πληρωμών 28,5% αλλά και για τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Για αυτές υπάρχει αύξηση για το εργαλείο της γειτονίας 4,9% και για τα υπόλοιπα προγράμματα αναλόγως. Ας πούμε για το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις 28% σε σύγκριση με πέρυσι. 78% Και για το ίστο μεθονούκλεα σε ελεκτικό Επίσης, σημαντικές αυξήσεις για τις πληρωμές. Κατά μέσο όρο κατά μέσο όρο σημαντική αύξηση. Για το εργαλείο γειτονίας 34,1%. Ευρωπαϊκό Assistant 33,7% 27,4% και για μικρότερα προγράμματα όπως την εξωτερική εγγύηση 78,1% Protection civile 44 Το instrument economics and building 35,2% και το ΑΔ 22%. Δηλαδή υπάρχουν αυξήσεις σημαντικές. Και για να είμαστε ρεαλιστές, η πρόταση αυτή θεωρούμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να θυμίσουμε ότι είναι έσχος ότι στο τμήμα αυτό 4 λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών πληρώθηκαν 1,7 εκατομμύρια μόνο και άρα θα συνεχίσουν τα προβλήματα και το 15 το 2016 πρέπει να έχει επιληθεί αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό λέω ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της Κομισιόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση διότι έβαλε περισσότερα χρήματα στις, για τις πληρωμές. Τώρα θα δούμε αν αυτά αρκούν, αλλά δεν ζητάμε και το αδύνατο. Τώρα για τις προτεραιότητες. Θέλω να δούμε τι φρονείτε κι εσείς, γιατί εγώ σκοπεύω κυρίως να ακούσω τις προτεραιότητές σας και να δω μετά αν μπορώ να κάνω ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό που να αναλαμβάνει τις ευθύνε που πρέπει να αναλαμβάνει και σέβεται τους συμβιβασμούς αλλά επίσης και προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες και επί των προτεραιοτήτων αυτών ήρθα να ακούσω τις ιδέες σας mm. και τις απόψεις σας. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φερνάντες σίγουρα θα σας πούνε πολλά οι ευρωβουλευτές μας. Οπότε ανοίγουμε τη συζήτηση με τον κύριο Πρέντα που είναι ο εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Φερνάντες πρώτα απ' όλα που ήρθε να ανταλλάξει απόψεις με τη δικιά μας την Επιτροπή. Θέλω επίσης να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για τη σημαντική αύξηση που έχουμε στο σχέδιο προπολογισμού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσον αφορά τις πιστώσεις υποχρέσεων και όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών στην κατηγορία 4 που έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπισμένος ότι προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να έχει το βάρος που θέλει να έχει στη διεθνή σκηνή πρέπει να πρικοδοτηθεί και αντίστοιχα με τις φιλοδοξίες της. Γι' αυτό και ο επιπλέον προπολογισμό, τα επιπλέον κονδύλια που προβλέπονται στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φρόσδεκτα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η αύξηση των πιστώσεων πληρωμών, χάρη στι οποίε θα υλοποιηθούν τα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πρωτοβουλίε για την σταθεροποίηση τη ειρήνη και άλλα προγράμματα τα οποία διακόπησαν για οικονομικούς λόγους. σκέφτομαι τις δραστηριότητε της Επιτροπής μας τον τελευταίο μήνα. Μια από τις σημαντικές μας προτεραιότητες είναι η γυτνίαση, τόσο προς Νότο όσο και προς Ανατολάς. Οπότε το ευρωπαϊκό μέσο για την γυτνίαση θα πρέπει να έχει αρκετούς πόρους ώστε να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τις χώρες που γειτονεύουν μαζί μας και που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Είναι επίση πολύ σημαντικό ο φετινό προπολογισμό να αντικατοπτρίζει και τι υποχρεώσει που έχουμε αναλάβει όσον αφορά την προστασία τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στι γείτονε χώρε όσο και πέρα από αυτέ. Έχω μια σύντομη ερώτηση προς τον κύριο Φερνάντες επίσης για την αντίδραση του Συμβουλίου. Έχει πάρει κανένα μήνυμα, κανένα σημάδι για το για την αύξηση που προβλέπεται στο σχέδιο προπολογισμού. Θα μπορέσουν να προχωρήσουν οι πληρωμές. Και επίσης, γενικά μιλώντας, ο τελικός προϋπολογισμός θα αντικατοπτρίζει την δέσμευσή μας υπέρ των γειτονικών μας χωρών, τόσο στο Νότο όσο και ανατολικά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον συνάδελφο Ζωζέ Μανουέλ Γκοζάλες <clears throat> για την έκθεσή του. Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες. Εγώ μιλάω και μέρου του σκιώδου συζητητή του κύριου Ζημανίσκη ο οποίο δεν μπόρεσε να έρθει εδώ σήμερα. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι πιστεύουμε πως θα ήταν χρήσιμο για τις επόμενες χρονιές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάζει το σχέδιο προϋπολογισμού πολύ πιο νωρίς με στη χρονιά ώστε να μπορούμε να αποφανθούμε και εμείς και να σχηματίσουμε άποψη ως Επιτροπή. Επίσης, ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να παίξει το ρόλο της ως παγκόσμιος παίκτη και να αντικατοπτρίζει τις γενικές προτεραιότητές μας. Τα κονδύλια δε οι πόροι πρέπει να συνάδουν με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε. Γι' αυτό και ο κύριος Φερνάντες εξάλλου θα εδώ να μας ακούσει. Συνεπώς, η ομάδα μου πιστεύει ότι ναι, είναι καλό που υπάρχει αυτή η αύξηση. 5,6% όσον αφορά την κατηγορία 4. Και τις πρώτες χρονιές στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αυτό πρέπει να φανεί. Επίσης συμφωνούμε για το ότι το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα να εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο για να προβάλλονται και ευρωπαϊκές αξίες. Όσον αφορά τώρα το μέσο για τη σταθερότητα και την ειρήνη, εδώ βλέπουμε ότι λαμβάνονται υπόψη δράσεις όπως είναι η αποστολή στο Σαχέλ Μαλή, στην Ουκρανία και επίσης και η αποστολή σχετική με τη Συριακή κρίση. Όμως δεν βλέπουμε να λαμβάνονται υπόψη η σύγκρουση, οι απειλές, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη Μεσόγειο. και κυρίως εξαιτία της κατάστασης στη Λιβύη. Για το λόγο αυτό η ομάδα μου θεωρεί ότι όσα έχουν συμπεριληφθεί δεν φτάνουν. Δεν θα φτάνουν για να μπορέσουμε με τις καθυστερημένες πληρωμές που έχουμε. Όσον αφορά την αύξηση 4,9 μονάδες όσον αφορά το μέσο γυπνίασης. Και εδώ πιστεύουμε ότι δεν αρκεί. Είναι σαφή, σαφές ότι η Συρία και η Ουκρανία αποτελούν προτεραιότητες, αλλά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν και που απορρέουν από τη Λιβύη πρέπει επίσης να λυθούν υπόψη και να υπάρξουν σχετικές προβλέψεις. Τέλος, πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη διαδικασία στη Μέση Ανατολή, παρόλο που βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ή δεν βρίσκεται, πιο σωστά, να στηρίξουμε δηλαδή την Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτά που αναφέρονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για μας δεν αρκούν για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ανάγκες, τα προγράμματα που προβλέπονται. Γι' αυτό και ζητάμε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών να το διορθώσει αυτό στον τελικό προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Φερνάντες. Επειδή δεν έχει ζητήσει κανένα άλλο συνάδελφο, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εμείς εγκρίναμε τις κατευθυντήριες γραμμές μας. Μετά ήρθε και έκανε την παρουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται για να λαμβάνει υπόψη τις δικές μας προτεραιότητες. Τώρα θα κάνει την ανάγνωση του το Συμβούλιο και στη συνέχεια το Κοινοβούλιο θα αποφανθεί Εμεί πολλές φορές επαναφέρουμε το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού έχει περάσει το Συμβούλιο από πάνω του. Ε, θα δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητε του Συμβουλίου. Ε, το Συμβούλιο έχει μια συνήθεια δεν να κάνει αυξήσει αλίμονο, αλλά κάνει πολλές περικοπές σε πολλές θέσει του προπολογισμού και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σχέδιο προπολογισμού για την πολιτική γειτονία προς Νότον και προς Ανατολάς. Έχουμε αύξηση για τον Νότο στις πληρωμές. Και είμαστε εντυπωσιακοί. 187,3% αύξηση των πληρωμών για τον Νότο και για την ανατολία 136,7% σε πληρωμές πάντα, όχι ανάληψη υποχρεώσεων. Αυτό τι σημαίνει ε, ότι είναι προτεραιότητα και θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για τις πληρωμές. Λοιπόν, από τη μια έχουμε την ανάληψη υποχρεώσεων, από την άλλη τις πληρωμές. Μα δεν είναι δυνατόν να ζητάμε τα θεσμικά όργανα να δώσουν τα επαρκή κονδύλια, αφού έχουν δεσμευτεί. Λογικό δεν είναι. Αφού τα έχουν τάξει θα πρέπει να τα ε, πληρώσουν κιόλας οι πληρωμές είναι μια απόρρια της ανάληψης υποχρεώσεων. Και ε, ε, όταν το, το Συμβούλιο εγκρίνει προπολογισμού, το κάνει με την ελπίδα ότι δεν θα τους εκτελέσουμε. Γιατί όταν έχει έρθει η ώρα της πληρωμής σημαίνει ότι ε, λειτουργούν οι πολιτικές και εκτελεί το προπολογισμό. Επιμένουμε εμείς αυτό, αλλά... Αν πήγαιναν όλα καλά, δεν θα χρειαζόταν να επιμένουμε. Επαναλαμβάνω, οι πληρωμές είναι λογική απόρρια και συνέπεια της ανάλυσης υποχρεώσεων. Τώρα, σε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού, το παρόν, για τις πληρωμές, το μέσο γειτονίας βλέπει μια αύξηση 34,1% και η ανάλυση υποχρεώσεων 4,9%. Εκεί θα πρέπει να είμαστε ε, υπεύθυνοι. Γιατί αν αυξήσουμε πάρα πολύ τις πιστός ανάληψης υποχρεώσεων, αν δεν ακολουθηθεί αυτό από τις απαραίτητες ε, πληρωμές, τότε διωγγώνουμε το πρόβλημα και δεν το λύνουμε. Για τη Μεσόγειο τώρα. Είναι σε άλλη κατηγορία, σε άλλο τίτλο, έτσι δεν είναι, που λέγεται τρία, ή το μέσο βελιξίας; 124 εκατομμύρια, πέρα από το περιθώριο δηλαδή, το αποθεματικό 124 εκατομμύρια για θέματα που έχουν να κάνουν με το άσυλο και τη μετανάστευση και την κρίση που γνωρίζουμε στη Μεσόγειο. Αυτό όμως είναι εκτός της ε, κατηγορίας 4 του τίτλου. Λοιπόν, θα ακούσω τις απόψεις σας, τη γνώμη σας και στη συνέχεια ξέρετε ότι πάντα δίνουμε μάχη κυρίως με το Συμβούλιο. Και όταν μιλώ για σεβασμό των ε, συμβιβασμών, των δεσμεύσεών μας, σημαίνει ότι ε, θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη, επαναλαμβάνω, γιατί έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις. Γιατί είναι όνειδος και ντροπή σκέτη στο 2004. Ε, ξέρετε πόσους στόχους έχουμε πληρώσει για ε, περίμενες πληρωμές. 1,7 εκατομμύρια. Ε, για καθυστέρηση πληρωμών και μόνο. Είναι μια κατάσταση αφόρητη και απαράδεκτη. Ε, ε, ευχαριστώ. Ελπίζω όσα σας είπαν τα μέλη της Επιτροπής μας να σας βοήθησαν. Εφόσον τα σημεία 5 και 6 αναβάλλονται, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να σταματήσουμε και στις 4 να επανέλθουμε με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.

μοντέλο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

πάρουν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

Vamos a, a reanudar. Λοιπόν, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Είμαστε στο σημείο 7, αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Θα συνεχίσουμε την εξέταση τροπολογιών της έκθεσης Κούκαν για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Έχουν κατατεθεί παρακαλώ 663 τροπολογίες. Mm. Καλός δείκτης λοιπόν της δραστηριότητας του Κοινοβουλίου και της πολυφωνίας. Θα δώσω μέσα το λόγο στον κύριο Κούκαν για να μοιραστεί μαζί μας ε, τις θέσεις του για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και τις ε, ιδέες του για να προχωρήσει η έκθεση. Έχετε το λόγο κύριε Κούκαν μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το τρομερό τους ενδιαφέρον στην έκθεση που κατέληξε σε 663 τροπολογίες οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες στην ανάγνωση. Εγώ έβαλα μερικές κυρίες ιδέες στην έκθεσή μου, θα τις αναφέρω σύντομα, τις έχω ξαναπεί βέβαια. Η πολιτική γειτονία πρέπει να είναι πιο στρατηγικών κατευθύνσεων υποστήριξη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι στο κέντρο της πολιτικής αυτής. Χρειαζόμαστε περισσότερο διαφοροποιημένες και ευλίγιστες ε, ε, προγράμματα. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τις πτυχές ασφαλείας της, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή ολοκλήρωση και την γειτονία με τους γείτονες. Χαίρομαι γιατί όλες αυτές οι ιδέες εγκρίθηκαν και εμπλουτίστηκαν από τις τροπολογίες. Μόνο μερικές από αυτές είναι κατά του γενικότερου τόνου του σχεδίου έκθεσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν ακόμη μια φορά για το ενδιαφέρον σας και για τη θετική σας προσέγγιση της έκθεσης. Καταρχήν θα ήθελα να επαναλάβω ότι ο στόχος μου είναι να είναι συνεπής και περιεκτική έκθεση χωρίς πολυλογίες. Και αυτό θα κάνω και με τις τροπολογίες και κατά τη σύνταξη των συμβιβαστικών. Θα ήθελα λοιπόν να πω εκ των προτέρων ότι θα υποστηρίξω τις γενικότερες ιδέες πολλών τροπολογιών, αλλά όχι με την ακριβή τους διατύπωση, αλλά με το νόημα χωρίς να χρησιμοποιήσω την ακριβή τους διατύπωση. Έχω ξαναπεί ότι η έκθεση αυτή πρέπει να αφορά την πολιτική γειτονία της Ένωσης και όχι συγκεκριμένες χώρες. Και αυτό δεν θα αναφέρω ποια είναι η κατάσταση σε συγκεκριμένες χώρες, στο κύριο τμήμα τουλάχιστον της έκθεσής μου. Επίσης θέλω να αφήσω περισσότερο χώρο για τις τροπολογίες που και αυτές ασχολούνται γενικότερα με την πολιτική γειτονία. Όσοι μετέφεραν τροπολογίε από άλλες εκθέσεις παρακαλώ να κατανοήσουν ότι δεν θα συμπεριληφθούν πλήρως αυτές. Τώρα για συγκεκριμένε τροπολογίε. Οι πρώτε 12 παράγραφοι είναι οι γενικές κατευθύνσει. και θα ήθελα αυτές να τις κρατήσω στον τόνο που είχα Υποστηρίζω όσες τροπολογίες τονίζουν το στρατηγικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Θα βρω άλλο μέρος για να βάλω τροπολογίες που μιλούν για θέματα διεθνούς δικαίου, περιφερειακής ολοκλήρωσης και αποφάσεις κυρίαρχων γειτονικών χωρών. Επίσης, οι τροπολογίες που ζητούν χωρισμό της ε, πολιτικής σε βόρειο και νότιο μέρος τις καταλαβαίνομαι, αλλά η θέση μου είναι να παραμείνει ενιαίο το πλαίσιο της ΕΠΓ και για να γίνει η διαφοροποίηση μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο. Όταν μιλάω για τη δημιουργία διαφορετικών επιπέδων συνεργασίας στην παράγραφο 5 εννοώ αυτή τη διαφοροποιημένη προσέγγιση την οποία προωθώ στο σύνολο της έκθεσης. Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να λέμε πιο σαφώς ποια είναι τα δικά μας συμφέροντα και όχι μόνο κοινέ προτεραιότητες κατά τον καθορισμό των στόχων της ΕΠΓ. Επίσης προτείνω πιο πολιτικού χαρακτήρα προγράμματα. Γι' αυτό ζητάω οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι να διατηρηθούν. Συμφωνώ με πολλούς από τους συναδέλφους που τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνέπεια μεταξύ της CSFP, CSDP και, και Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι αυτά τα θέματα ήδη αναφέρονται στην παράγραφο 21, άμα τη διαβάσετε προσεκτικά στην παράγραφο 8 όταν μιλάμε για δωρητάς και το συντονισμό τους είδα ότι πολλές τροπολογίες αναφέρουν το MSCI το συντονισμό επενδύσεων για τη Μεσόγειο δηλαδή. Αυτό θα το ξαναδώ αργότερα. Στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης γίνεται λόγος για αναμόρφωση της ΕΠΓ και οι περισσότερες τροπολογίες εκεί είναι τροπολογίες που τις δέχομαι εκτός από εκείνες που αναφέρουν την προσέγγιση λιγότερα για λιγότερα. Δεν βλέπω καμία ανάγκη να τις προωθήσω αυτές τις ιδέες. Παράγραφος 13 αφορά διαφορετικές έννοιες της διεύρυνσης και της πολιτικής κοινωνίας καθώς και τα άρθρα της συνθήκης θέλω να αναφέρονται και τα δύο αυτά θέματα. Στην υποστήριξη για δημοκρατία και θεσμικό capacity building επίσης δεν βλέπω προβλήματα με τις τροπολογίες. Τις περισσότερες προσθήκες που αφορούν δικαιώματα και ελευθερίες θα τις συμπεριλάβω καθώς και εκείνες που τονίζουν την καλή διακυβέρνηση και την οικοδόμηση κρατών. Στα πλαίσια της ΕΠΟΓΟ επίσης νομίζω ότι καλό είναι εκεί να αναφέρονται και τα δικαιώματα γυναικών και παιδών που αναφέρουν πολλές τροπολογίες. Στο τμήμα για τη διαφοροποίηση και τους όρους επίσης δεν βλέπω φοβερά προβλήματα. Στην παράγραφο 18 θα ήθελα να παραμείνω τους όρους που τονίζουν την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και των αξιών της Ένωσης καθώς και της προσέγγισης παραπάνω για παραπάνω. Τώρα για την ασφάλεια, σημαντικό τμήμα της έκθεσης. Δέχομαι τις τροπολογίες που προσθέτουν την παραπομπή στο οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία, στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κρίσεων από την Ένωση και τη μεγαλύτερη συνέπεια με την πολιτική ασφαλείας η στρατηγική ασφαλεία. Οι τροπολογίες που αφορούν την επίλυση παγωμένων διαφορών επίσης νομίζω πρέπει να ε, έχουν χωριστή παράγραφο. Αλλά θα ήθελα να παραλείψω από το τμήμα αυτό τις παραπομπές στην μετανάστευση γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ευρύτερο από τα θέματα της ασφαλείας. Επίσης δεν θα ήθελα να συμπεριληφθούν αναφορές σε συγκεκριμένες αποστολές και επιχειρήσεις της Ένωσης. Ε, όσο για την περιφερειακή συνεργασία και τους γείτονες των γειτόνων, ε, ακούγονται πολλές ιδέες από τις τροπολογίες και θα προσπαθήσω να τις συμπεριλάβω στις συμβιβαστικές. Αλλά θα προσπαθήσω να αποφύγω αναφορά συγκεκριμένων χωρών ή περιφερειών χωρών στην πολιτική γειτονία. Όσο για τις κυρίαρχες επιλογές ορισμένων χωρών, εδώ θα στηρίξω τις τροπολογίες αυτές. Τελικό τμήμα. Οι στόχοι και τα εργαλεία της πολιτικής αυτής, όπου ήθελα να ταυτίσω τις προτεραιότητες της συνεργασίας κλπ. Δεν θέλω να είμαι πολύ περιοριστικός εδώ σε αυτό το τμήμα, αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσω να μην δοθεί η εντύπωση ότι όλα είναι προτεραιότητα. Γιατί δεν είναι. Γι' αυτό θα συζητήσω με προσοχή με τους σκιώδεις αυτές τις τροπολογίες και θα προτείνω συμβιβαστικές. Ιδιαίτερα ως προς τα άρθρα 31 και 32 σημεία. Επίσης γνωρίζω ότι το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας αλλά και της μετανάστευσης είναι λεπτό και θα προσπαθήσω να τα ταιριάξω και εκεί. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τον ενδιαφέρον τους. Θα παραμείνω σε στενή επαφή μαζί τους με τους κοιόδης για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές που θα ετοιμαστούν πολύ γρήγορα και προσβλέπω στην συζήτηση είμαι ανοιχτός σε συντάσεις και σχόλιά σας. Τέλος, επειδή 663 τροπολογίες είναι μεγάλος αριθμός, δεν μπορώ να τους ικανοποιήσω μάλλον όλους και ίσως να απογοητευτούν μερικοί. Επίσης θα ήθελα να σας ζητήσω να μην κάνετε πολύ πολύπλοκες και καινούργιες διατυπώσεις των ίδιων πραγμάτων γιατί δεν θα χωρέσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούκαν. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χάουικ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ του συναδέλφου Άντι Κριστέα που είναι ε, σκιώδης εισηγητής στην έκθεση του κυρίου Κούκαν εξ ονόματος της ομάδας μου και όλων των υπολείπων θέλω να το ευχαριστήσουμε κάνει τρομερή δουλειά, είναι πάρα πολύ εξέχων ευρωβουλευτής και ε, εξαιρετικό τέλεχος και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Ε, τι λέει λοιπόν η δική μας πολιτική ομάδα. Αυτό το γεγονός ότι είναι 663 τροπολογίες δείχνει πόσο πολύ ενδιαφέρει ε, τον κόσμο αυτή η πολιτική γειτονία και πόσοι βουλευτές ενδιαφέρονται να επιτύχει και να δώσει καρπούς. Λέει ο εισηγητής ότι είναι συγκλίνουσε σε μεγάλο βαθμό οι τροπολογίες, δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, από τη μία τροπολογία στην άλλη. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ε, στις διαπραγματεύσεις και στις συμβαστικές τροπολογίες που θα φέρει ο εισηγητής θα είναι μια πολύ γερή βάση για συνένεση. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τα βασικά στοιχεία ε, των Σοσιαλδημοκρατών και που θέλει και ο κύριος Κριστέα να μπουν στην έκθεση και ξέρω πολύ καλά ότι τα κατανοεί ο εισηγητής. Εμείς δεν έχουμε διαφορετικές αξίες ή διαφορετικά στάνταρ και αξίες και αρχές που λέμε ότι είναι καλές στην την Ευρώπη είναι εξίσου καλές και για τους γειτονές μας. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις δηλαδή, ε, ούτε θα περιορίσουμε τις αρχές και τις αξίες μας. Δεν υπάρχει τέτοιο, είναι ψευτοδήλημα αυτό ε, και θα πρέπει να το ξέρουμε. Επίσης θέλουμε μεγαλύτερη σύγκληση ανάμεσα στην πολιτική ε, γειτονία στην ΚΕΠΑ και την ΕΠΑ. Δεν είναι διαφορετικές πολιτικές, είναι πολιτικές εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Θα πρέπει να ε, αξιοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στην εξωτερική μας πολιτική για να προωθούμε αυτές τις δράσεις και προς τις γειτονικές μας χώρες. Και γι' αυτό ε, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να θεωρούνται διακριτές αυτές οι πολιτικές εξεχωριστές μεταξύ τους. Θα πρέπει να δοθεί ε, έμφαση στη ρίζα των δεινών, ορισμένων προβλημάτων. Σημείωσα αυτό που είπε ο κύριο Κούκαν για τη μετανάστευση, για τη Μεσόγειο. Είναι δύσκολο βέβαια να κρατηθούν εκτός της έκθεσης, για να είμαι ε, ελπίζω να το μελετήσετε και να προτείνετε κάποιους λογικούς συμβιβασμούς και δίκαιους. Αλλά πραγματικά σας συγκετεύουμε να τα κοιτάξετε αυτά τα θέματα. Είναι τεράστια τα προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπίζουμε όχι μόνο τα συμπτώματα αλλά και τα αίτια. Και δεν είναι μόνο η μετανάστευση. Η ομάδα μας επίσης προσπαθεί να εξασφαλίσει την πληροφόρηση, την επικοινωνία, την προβολή μας. Δεν είναι τα αρκετά ορατές οι πολιτικές μας. Ιδιαίτερα στην πολιτική γειτονία. Έχουμε κάποιες καλές πολιτικές, αλλά δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να τις προβάλλουμε, στο να τις πουλάμε εντό εισαγωγικών. Ε, δεν τα ξέρουν όλα αυτά που κάνουμε στις ε, γειτονικέ μας χώρες. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις σε αυτό το τομέα. Επόμενο θέμα. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η διαδικασία αυτής της γειτονίας παραμένει ανοιχτή για τις χώρες που θέλουν να ενταχθούν. Είναι δύσκολο να το πεις αυτό τον καιρό που υπάρχει αυτή η λεγόμενη κόποση από τις διευρύνσεις και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, άνδρες και γυναίκες προσπαθούν ε, να απομακρυνθούν από τη διεύρυνση. Εμεί είμαστε κοινοβούλιο, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Φυσικά δεν μπορεί αύριο να γίνει η διεύρυνση για ορισμένε από τις χώρες, αλλά να μην τους κλείσουμε την πόρτα Υπάρχουν χώρες που θέλουν να μπουν στον ευρωπαϊκό δρόμο και υπάρχει αυτή η δυνατότητα της γειτονία. Είναι σημαντικό και αυτό το στοιχείο της έκθεσης και θέλουμε να το πούμε. Να πω και κάτι προσωπικό τώρα για τις δικές μου τροπολογίες. Όλα αυτά που έλεγα τώρα ήταν του Κριστέα πρέπει να πω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για τη δέσμευση και την προσήλωσή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, γιατί υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να μας παρεξηγήσουν. Ε, σε ό,τι μας αφορά λοιπόν εμάς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και θέλω να έχουμε καλύτερες και πάλι επιδόσεις ε, ε, απέναντι στα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών, συνεργαζόμενοι μαζί τους, όταν έχουμε χώρες με, μετάβαση, πώς μπορούμε ε, να βοηθήσουμε τον κόσμο που είναι εκτός του πολιτικού γίγνεσθε να ενταχθεί σε αυτό, τα κινήματα ας πούμε. Το έχουμε συζητήσει και αυτό στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και ε, σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη, ενδεχομένως και για την Ουκρανία Ξέρω ότι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις αναχώρα και να προτείνουμε στην έκθεση, αλλά πραγματικά να βοηθήσουμε όχι μόνο την πολιτική τάξη εκεί και το πολιτικό σύστημα, αλλά περισσότερο τους πολίτες να συμμετέχουν. Για τι δικέ μου τροπολογίε ακόμη, θέλω να επιστήσω την προσοχή στο, στο εξή. Πολλοί εδώ μέσα, στην Επιτροπή μα και στο Κοινοβούλιο, διαρριγνύουν τα ημάτια του για την ΚΕΠΑ, για την ΕΠΑ και τελικά ε, στη γειτονία αποτυγχάνουμε. Βεβαίως έχουμε στόχους για την ΚΕΠΑ και με άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά όταν δεν τα κάνουμε στη γειτονιά μας αυτά, πώς μπορούμε να τα πρεσβεύουμε ανά την υφήλη, όταν δεν έχουμε την πολιτική βούληση, τα μέσα ή την ενότητα για να συμφωνήσουμε για πολύ δύσκολες και κρίσιμες καταστάσεις. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η πολιτική γειτονία ε, είναι μια δοκιμή ε, με βάση την οποία κρίνεται η γενικότερη εξωτερική πολιτική της Ένωσης, είτε είναι ασφάλειας και άμυνας, είτε είναι η ΚΕΠΑ. Οπότε ε, ελπίζω να βοήθησαν αυτά που είπα στη σημερινή συζήτηση. Προσβλέπουμε πάρα πολύ στη συνεργασία μας με τον κύριο Κούκαν στις επόμενες συνεδριάσεις των σκιωδών και να δούμε και τις συμβαστικές. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι επικοδομητικές και η έκθεση θα είναι πάρα πολύ καλή τελικά. Με πολύ μεγάλη συνένεση. Ευχαριστώ πολύ. Gracias, señor Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε ο Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Φυσικά και υπάρχει ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία και είναι σημαντικό αυτό και το διαπιστώνουμε και από τις πολλές τροπολογίες. Αυτό δείχνει τον επερχόμενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τι βαθμό θα είμαστε σημαντικοί, αποτελεσματικοί και σε τι βαθμό θα τηρήσουμε τις δικές μας τις υποχρεώσεις προκειμένου να έχουμε σταθερότητα και στις δικές μας χώρες και στις δικές μας γείτονες χώρες. Ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Κούκαν. Ήταν πολύ σημαντικά τόσα μας είπατε τροφή για σκέψη προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποιες αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε συμβιβασμού στη συνέχεια. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το σωστό πλαίσιο για την κατάσταση αυτή. Συμμεριζόμαστε την απόψή σας για το ότι αν συγκεντρωθούμε πολύ σε επιμέρους χώρες θα δυσκολευτούμε να δούμε το σύνολο. Σίγουρα όμως υπάρχουν και πτυχές που είναι πολύ σημαντικές και χωρίς να τις αναφέρουμε δεν καταφέρουμε να καθορίσουμε τους μελλοντικού μας στόχους. Γι' αυτό και η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών θέλει το εξή. Η κατάσταση ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γνωστή. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, καταλαβαίνουμε τι γίνεται με τη ρωσική επίθεση στην εδαφική κυριότητα της Ουκρανίας, κατάσταση που κλιμακώνεται. Η κατάσταση στην Ουκρανία θα καθορίσει τι θα γίνει και σε άλλες χώρες ανατολικά των συνόρων μας. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα. Δεύτερο, η τροπολογία 71. Η Γενική Αρχή που πρέπει να υπάρχει στο συμβιβασμό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την κυριαρχία των χωρών που είναι γειτονέ μας και εταίροι μας. Είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς και για μας. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται ανεξάρτητα. Και τώρα πάμε νότια της Ευρώπης, στην νότια διάσταση της πολιτικής γειτονίας. Επικεντρωνόμαστε στη σχέση της ε, σταθερότητας στις χώρες που βρίσκονται ενωτίως ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις συγκρούσεις που υπάρχουν εκεί και αυτό το συνδέουμε με τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Σίγουρα οι ρίζες της μετανάστευσης μπορεί να είναι η οικονομική διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου. Μακροπρόθεσμα αυτό θα καθορίσει την κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι τα πρόσφατα προβλήματα απορρέουν από τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα και που δεν έχουν λυθεί στις περιοχές εκείνες από όπου μας έρχονται οι μετανάστες. Η πολιτική λοιπόν η ευρωπαϊκή γειτονία θα πρέπει να την αναφέρει αυτή την πτυχή. Οι εμφύλοι πόλεμοι και άλλες συγκρούσεις που συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή ακριβώς του κόσμου. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, κάτι που για μας έχει μεγάλη σημασία και το αναφέρουμε στη τροπολογία μας 323. Σωστή προσέγγιση όσον αφορά τους κοινωνικούς στόχους ή τέλο πάντων στόχους που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ευθύνη. Πολύ συχνά αναφερόμαστε στη δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Νότος είναι η ελευθερία των χριστιανών, των κοινοτήτων των χριστιανών. Άμα θέλουμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να νιώθει υπεύθυνη για όλες τις μειονότητες ε, που βρίσκονται σε δυσκολία, δεν θα τα καταφέρουμε αν δεν δεχτούμε ότι τέτοιες χριστιανικές κοινότητες επίσης πρέπει να προστατευτούν, είναι ευάλωτες δηλαδή είναι δικιά μας ευθύνη εξαιτίας των αρχών μας, της ιστορίας μας, αλλά και εξαιτίας των προσδοκιών εκατομμυρίων Ευρωπαίων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους. Επίσης, πρέπει να προσπαθήσουμε αυτές οι πτυχές τα θέματα τα οποία σας ανέφερα να συμπεριληφθούν και στους συμβασμούς. Ελπίζω το τελικό κείμενο να αντικατοπτρίζει την άποψη όχι μόνο της δικιάς μας της πολιτικής ομάδας αλλά και ολόκληρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριο Στραφίτσιος. Έχουμε πολλούς βέβαια ομιλητές. Δύο λεπτά παρακαλώ ο καθένας για να προλάβουμε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, ο κύριος θα είμαι σύντομος και συγκεκριμένος για κάποια θέματα που μας απασχολούν όλους. Ο κύριος Κούκαν πράγματι ανέλαβε πολύ σημαντικό έργο όσον αφορά τις χώρες που γειτονεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μεγάλες, είναι διαφορετικές, έχουν διαφορετικά προβλήματα και είναι περίπου το μισό του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε Κάθε φορά που μιλάμε για αυτά τα θέματα, να δεχτούμε ότι οι χώρες αυτές είναι διαφορετικές και άρα πρέπει να τις διαφοροποιήσουμε και όχι μόνο μεταξύ νότου και ανατολικής πλευράς. Εμείς θέλουμε τις χώρες αυτές να τις δούμε σαν εταίρους μας, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιες βασικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους, γεωγραφικά αν μη τι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν αυτό θα το τόνιζα πολύ. Η οικοδόμηση ικανοτήτων. Θέλω να ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους να συμφωνήσουν με αυτό το θέμα και να επιτρέψουν σε που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία, με την οικοδόμηση ικανοτήτων, να έρθουν με νέες ιδέες. Επίσης προτιμάω να μιλάω για more for more, περισσότερα για περισσότερα, παρά για less for less. Το αντίθετο δηλαδή, λιγότερα για λιγότερα. Έπειτα, νωρίτερα αναφερθήκαμε στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τους γείτονές μας. Είναι κάτι διαφορετικό από την αναπτυξιακή βοήθεια προς τρίτες χώρες. Η πολιτική γειτονία λοιπόν πρέπει να αποτελεί ένα μέσο όθησης. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τις ικανότητες του συναδέλφου του κ. Κούκαν, είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε πάρα πολύ καλές συμβαστικές προτάσεις. Προσβλέπω σε συνεργασία μαζί του. Ο κύριος Σόλτς, ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τους προλαλήσαντες. Έζησε το μικρόφωνο όμως του κυρίου Σόλτσβαρκ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κούκαν για την προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτή τη τεράστια πρόκληση και την αναθεώρηση, την αναδιατύπωση. Θέλω να θυμίσω κάτι καταρχήν. Είχαμε πολύ επικοδομητική και καρποφόρα συζήτηση στο έγγραφο εργασία. Την πρώτη φορά που το παρουσίασε ο εισηγητή και περιέγραψε, αν θυμάστε τότε, του στόχου και τα μέσα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθούν, να αναθεωρηθούν με βάση μια πάρα πολύ κριτική ανάλυση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων. Και συμφωνούμε όλοι εδώ, είναι κοινή αντίληψη ότι πρέπει να ξαναδούμε αυτό το θέμα της γειτονίας και προς Ανατολάς και προς Νότον. Για να δούμε ποιοι είναι λοιπόν οι πολιτικοί στόχοι, εξακολουθεί να ισχύει και το αυτό και το έγγραφο εργασίας και η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης νομίζω όμως ε, δεν το λέει τόσο ρητά. Και ποιο είναι αυτό. Θα πρέπει να έχουμε στρατηγικούς στόχους αλλά και πολιτικό όραμα που να συνδέεται με αυτούς. Τι σημαίνει αυτό. Το πολιτικό όραμα έχει ε, χρειάζεται διαφοροποίηση, ευελιξία, εστίαση, ε, ίδια ευθύνη και προβολή. Και αυτό σε διαφορετικό βαθμό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός και για τις χώρες γειτονίας αφετέρου. Και αυτά θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρα διαχωρισμένα. Και έχουμε να ρωτήσω το εξής, για να είμαστε και πιο συνεκτικοί στην πολιτική μας. Γι' αυτό κάναμε και τροπολογίες για την Ανατολή και για τον Νότο, επαναλαμβάνω. Πώς λοιπόν μπορεί η δράση, κοινωνική, η οικονομική, η περιβαλλοντική, η δράση στα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες που είναι τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Εμείς προσπαθήσαμε ως ομάδα ε, να κάνουμε ε, τροπολογίες όπως είναι οι 10, 16, 36 και 70 για να δούμε πώς θα επιφέρουμε μεγαλύτερη συνοχή. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε μόνο πολιτική γειτονία γενικά και αόριστα. Αυτό έχει και πτυχές και συγκεκριμένες επιπτώσεις σε άλλους τομείς της πολιτικής, κοινωνική, πολιτική, οικονομική, συνεργασία, αναπτυξιακή και πάει λέγοντας. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή. Ελπίζω να καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς για μια καλή έκθεση, για μια καλή αναθεώρηση της πολιτικής αυτής. Ευχαριστώ. Έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Ο κύριος Μέσαρικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αρχίσω ευχαριστώντας και συγχαίροντας τον εισηγητή. Είναι από τα δυσκολότερα πράγματα να προσπαθήσει κανείς να συνδυάσει τόσο πολλά θέματα όσο αυτά που θίγει η ΕΠΓ. Υπάρχουν θέματα επί των οποίων συμφωνούμε και εμείς απολύτως και τροπολογίες Επίσης, εγώ προσωπικά υποστηρίζω ας πούμε την ιδέα των ειδικών απεσταλμένων ακόμη και αν μερικοί διαφωνούν. Τώρα, υπάρχουν δύο θέματα που θα ήθελα να θίξω. Το ένα είναι η αρχή more for more. Συμφωνήσαμε ως ομάδα ότι η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα και ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι όροι για την εφαρμογή της όπως λέει και η παράγραφος 18 και ότι μπορεί αυτό να πετύχει το στόχο του αλλά παρόλα αυτά και η ιδέα less for less δεν είναι καταστροφική. Απλώς αν δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε όπως πρέπει το more for more ή υποχωρήσουν ορισμένοι γείτονες, τότε δεν θα έχουμε κανέναν τρόπο αντιμετώπισης. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της ασυνεπούς, μιας ασυνεπούς εφαρμογής του More for More. Επίσης, κατανοούμε τη διαφοροποίηση που γίνεται για το σύνολο της ΕΠΓΟ και είναι λογική, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν περιφερειακά στοιχεία που ενδιαφέρουν την Ένωση ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο και ότι πρέπει αυτά να αναθεωρηθούν και να επανεξεταστούν γιατί φαίνεται ότι μέχρι τώρα οι συνεννοήσεις για τη Μεσόγειο είναι τελείως καταστροφικές και έχουν τελείως καταστροφικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Σαφχάουζερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρία πράγματα για την πολιτική διεύρυνση που θα πρέπει περισσότερο να αναδειχθούν. Πρώτον, η κυριαρχία η κρατική κυριαρχία, εθνική κυριαρχία των χωρών, το λεγόμενο κοινοτικό και εκτιμένο ή ενωσιακό δεν θα πρέπει να αντιτίθεται σε αυτή την εθνική κυριαρχία που ε, συνδέεται με την ελευθερία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να πετύχει διεύρυνση. Κατά τα άλλα, το έγγραφο της κυρίας Μογκερίνη έρχεται να υπογραμμίσει πολύ συχνά ότι δεν έχουμε δώσει ιδιαίτερη αρκετή προσοχή στην κυριαρχία των διαφόρων κρατών. Και έχουμε λίγο εμπειριελιστική τακτική και συμπεριφορά. Δεύτερον, θα πρέπει να μην κόβουμε τι γέφυρε. Εγώ κατάγομαι από την Αλσατία. Η Αλσατία 700 χρόνια ε, ήταν γερμανική και στη συνέχεια με τον Λουδοβίκο το 14ο ε, ήρθε στη Γαλλία. Δηλαδή είναι τμήμα και της Γαλλίας που έχει ένα γερμανικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι και ισχύ τη. Και αν έπρεπε να μας πούνε, διαλέξτε ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, όταν χρειάστηκε να μας το πούνε αυτό, οδηγηθήκαμε σε δύο παγκοσμιου πολέμους. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τις γέφυρε και μιλώ για την Ανατολική Ουκρανία. Ο Στάλιν αυτές τις περιφέρειες τις έβαλε στην Ουκρανία, διότι, όπω έλεγα σε ένα συνάδελφο, ε, είχε πρόβλημα με τη Γαλλική εκεί και τι δυτικέ περιοχές και θα πρέπει να ε, ε, κατανοήσουμε και να διατηρήσουμε την ιδιαιτερότητα αυτών των περιοχών σε όλη την πολιτική γειτονία θα πρέπει να αρνηθούμε αυτή την ε, σύγκρουση ε, Ανατολής δύση. Δύο παγκοσμίου πολέμου είχαμε εξαιτία αυτού, να μην προετοιμάσουμε και ένα τρίτο τώρα. Ταυτόχρονα να σταματήσουμε τον πόλεμο και να ε, επιβάλλουμε, για να επιβάλλουμε τη δημοκρατία. Δεν γίνεται με πόλεμο αυτό. Γίνεται βήμα-βήμα. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο δημοκρατία. Αυτοί που θέλουν να επιβάλλουν το μοναδικό μοντέλο τη δημοκρατία, αν κοιτάξουμε τι γίνεται στι χώρε του δεν είναι γνήσιοι δημοκράτε αυτή λογική ότι κάνω πόλεμο για να επιβάλλω την ειρήνη ή τη δημοκρατία είναι τελείως ε, απολυταρχική, ολοκληρωτική και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τη δεχτούμε, την αποκρούμε αναφανδών. Αυτά τα τρία είχα να πω και ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πλένκοβιτς. Ε, ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Περμούη. Ε, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω για τις καλές εξηγήσεις του κύριο Κούκαν. Μας εξήγησε πολύ καλά τις ε, τροπολογίες και τις ομαδοποίησε. Θα ήθελα εγώ να πω το εξής. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το timing. Δηλαδή, αμέσως μετά τη Σύνοδο κορυφή της Ρήγα, έχουμε αυτή την έκθεση και συζητούμε. Ε, είναι θετική, ε, παρόλο που βλέπει με ε, κριτικό μάτι τις χώρες γειτονίας και κάνει διαφοροποίησεις ανάλογα με τις χώρες. Επίσης, η πολιτική γειτονίας δοκιμάζεται και ως προς τη λειτουργία της και προς την αξιοπρέπειά της και προς την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς. Θα ήθελα αυτό να μπει ως ιδέα στην αρχή της έκθεσης, ως προήμια, Για το διεθνές δίκαιο τώρα και κατά πόσο γίνεται αυτό σεβαστό. Δηλαδή, ότι δεν θα πρέπει ορισμένες αρχές και αξίες να επιβάλλονται με τρόπο επιθετικό. Εδώ συζητούμε για την Επιτροπή Γειτονίας και υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας η οποία αυτό τον καιρό αναθεωρείται και ε, μέχρι το 2016 θα έχει ολοκληρωθεί αυτή. θα έχουμε μια νέα διαμόρφωση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, όλα τα εργαλεία που έχουν αποδειχθεί χρήσιμα στην ε, πολιτική διεύρυνση. Τι εννοώ, την οικονομική διακυβέρνηση για παράδειγμα. Ή ε, αυτό το εργαλείο μπορούμε να το μεταφέρουμε ε, στην ε, Ανατολική και στη γενικότερη γειτονία ή ε, να είναι υγιή τα δημόσια οικονομικά μιας χώρας. Αυτά είναι θετικά παραδείγματα που πρέπει να μεταφερθούν. Και ελπίζω και ο Επίτροπος Χάν στα τέλη του έτους να προτείνει μια στρατηγική καλύτερη και ευρύτερη. Κατά τα άλλα ευχαριστώ πολύ τον συγητή και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βερτέλγης τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, κύριο Σπέτελε. Εδώ συζητάμε για μια πολύ σημαντική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι η έκθεση του κ. Κούκαρα αντικατοπτρίζει τις πραγματικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις χώρες με τις οποίες γειτονεύουμε. Η κατάσταση είναι λιγότερο ρομαντική από τότε που ξεκινήσαμε να προβληματιζόμαστε για το πώς θα αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με τις γείτονες χώρες. Σήμερα υπάρχει αποσταθεροποίηση, κατακαιρματισμός και είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτό για μας. Το ερώτημα είναι πώς κάνουμε τα πράγματα. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε τις αρχές μας και τις αξίες μας. Αυτό λέμε τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση όμως σήμερα είναι διαφορετική. Μιλάμε για διαφοροποίηση. Δεν μιλάμε για την εφαρμογή των δικών μας αρχών και αξιών. Η έκθεση Κούκαν λοιπόν πιστεύω ότι αποτελεί ένα έγγραφο το οποίο θέλει να ενισχυθούν οι αξίες μας όσο γίνεται περισσότερο βάσει των συνθήκων. Έχουμε όμως διαφοροποίηση πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι περισσότερες χώρες που βρίσκονται κοντά μας είναι χώρες που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εκδημοκρατισμό τους. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να υπογραμμίζουμε περισσότερο τα ρεαλιστικά στοιχεία μιας καλής διακυβέρνησης. Έχουμε πολλά προβλήματα λοιπόν με τις γείτονες χώρες, επειδή η καλή διακυβέρνηση δεν έχει ε, πάρει σάρκα και ως εκεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού. Εγώ θέλω να συνεργαστώ ευχαρίστω με όποιον θέλει να συνεργαστεί μαζί μας εφόσον συμμεριζόμαστε τα ίδια συμφέροντα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Θέλω να, και εγώ να πάρω το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κούκαν. Στην ε, γειτονία όμως νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που μας απασχολούν. Γιατί, Γιατί δεν πιστεύω ότι μπορούμε να ξεχνάμε αδικίες που αντιμετωπίζουν οι Σαχαραοί, οι Παλαιστίνοι ή άλλες πολύ σοβαρές καταστάσεις όπως είναι εκείνες που βλέπουμε σήμερα στη Συρία και τη Λιβύη. Γι' αυτό και εμείς έχουμε υποβάλει τροπολογίες και θα σας αναφέρω κάποιες από αυτές. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια βιώσιμη κατάσταση στην περιοχή και αναφερόμαστε στη Συρία. Ο Στάφα Τεμαστούρο που είναι ειδικό απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να έχει αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε ότι ορισμένες χώρες βοηθούν με εξοπλισμό. Όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική, τα βλέπουμε και στη Λιβύη και αλλού και στη Συρία, τις εξωτερικές παρεμβάσεις. Πρέπει να καταγγείλουμε λοιπόν το ρόλο που παίζουν χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Σεντική Αραβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Παλαιστίνη και εκεί είναι ζωτική σημασία. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή και θα υπάρχει αν υπάρχει και στην Παλαιστίνη. Εγώ έρχομαι από την Ισπανία. Και θα έλεγα γι' αυτό ακριβώς ότι πρέπει να σταματήσει η κατοχή ε, στην Δυτική Σαχάρα και το Μαρόκο να συμμορφωθεί για να αποπικραπηθεί η περιοχή. Μια μεγιά μου επόμενος ομιλητής. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Κούκαν. Συμφωνούμε με τις βασικές γραμμές τις κύριες γραμμές της έκθεσής του και τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή του. Σίγουρα έχει πολλή δουλειά με τις τροπολογίες, αλλά με την εμπειρία που έχει και τις ικανότητές του θα τα καταφέρει. Παρόλο που είναι τόσες πολλές οι τροπολογίες. Θέλω να αναφέρω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, και δεν νομίζω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή. Πρέπει να έχουμε μια ενία πολιτική όσον αφορά την γειτονία με δύο διαστάσεις. Αλλά δεν μπορούμε όπως λένε ορισμένοι ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές πολιτικές γειτονίες ανάλογα με τη χώρα. Στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Γειτονία αναφέρονται δύο διαστάσεις και όχι διαφορετικές πολιτικές, επειδή ορισμένες χώρες βρίσκονται ανατολικά και άλλες νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, η διαφοροποίηση πιστεύω ότι είναι αναγκαία. Σίγουρα tailor-made, όπως λέει ο κύριος Κούκαν, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα, τις φιλοδοξίες αλλά και τις ανάγκες των χωρών και να έχουν συμφωνηθεί όλα αυτά με τις ίδιες τις χώρες. Θέλουμε να έχουμε ρεαλιστική πολιτική που να μην είναι μια χήμερα και που να τις έχουμε συμφωνήσει με τις ενδιαφερόμενες χώρες και για τις χώρες ανατολικά της Ευρώπης και για τις χώρες νοτίως της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε τη... και τη Βαρκελόνη που να... δεν πρέπει να γίνεται κάθε 8 χρόνια όπως έγινε τελευταία. Και υπάρχει και κάτι άλλο και θα τελειώσω με αυτό. Η σημασία που έχει ασφάλεια, το είπε και ο κύριος Κούκαν. Δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε στην πολιτική μας γειτονία, ούτε και το θέμα της μετανάστευσης μπορούμε να παραβλέψουμε. Ο κύριος Κούκαν νομίζω ότι αντιμετωπίζει αυτό το θέμα τις μεταναστευτικές ροές, την ε, αναλογία με την οποία θα τις δεχόμαστε Πρέπει να υπάρχει τάξη στις μεταναστευτικές αυτές ροές, να μην υπάρχουν παρατυπίες. Είναι μια πτυχή για την οποία πρέπει να κάνουμε μια παραπάνω προσπάθεια και να φροντίσουμε να υπάρχει συνεργασία εκατέρωθεν της Μεσογείου. Σωστά στηρίζει την αρχή του περισσότερα και περισσότερα ο εισηγητής πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και όχι κυρώσει. Συνεπώς, πολύ σωστή αυτή η ιδέα του περισσότερα και περισσότερα και να βοηθήσουμε τις χώρες που κάνουν μεταρρυθμίσει, λαμβάνοντα υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα και την πρόοδό τους όμως. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κούκαν. Thank you, Mr. Chairman. Uh, very brief. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και τους μεμονωμένους συνάδελφους που έλαβαν το λόγο στη συζήτηση αυτή. Με ενθάρρυναν αυτά που άκουσα, γιατί ήδη είδα ότι όλοι επιθυμούν να συνεισφέρουν και μάλιστα θετικά για να έχουμε μια καλή έκθεση που θα αντανακλά όσο γίνεται περισσότερο το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα καταδεικνύει πόσο αποφασισμένο είναι να έχει συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερα στην αρχή, χάρη στο γεγονός ή εξαιτία του γεγονότος ότι υπάρχουν τόσο πολλές τροπολογίες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμπεριληφθούν όλες ε, στις συμβαστικές. Ε, τα είπαν κάποιοι συνάδελφοι και ο κύριος Σόλτ και ο κύριος Σέμερης. Υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται περισσότερη συζήτηση και θα το κάνουμε ε, στις συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών εν ώψη του συμβιβασμού. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και για κάτι δύο διμερείς συναντήσεις. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη συζήτηση για να καταλήξουμε. Σε ορισμένε περιπτώσεις Μπορεί να υπάρξει δυσκολία να ικανοποιηθούν όλες οι τροπολογίες, το είπα στην αρχή. Αν αρχίσουμε τώρα να διηλίζουμε τον κόνοπα ε, ως προς την εσωτερική πολιτική κατάσταση κάποιες χώρες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε κάτι, πώς να το πω, συνεκτικό. Γιατί χρειαζόμαστε μια σύντομη έκθεση και στην έκτασή της. Σας ευχαριστώ, σας ζητώ την κατανόησή σας και την ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις για να καταλήξουμε σε όσο γίνεται μεγαλύτερη συμφωνία για την έκθεση αυτή, γιατί το αξίζει πραγματικά και έχει σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούκαν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε στην έκτακτη συνεδρία στο Στρασβούργο στις 11 Ιουνίου. Και τώρα έχουμε την επόμενη συνεδρίαση που είναι και κλεισμένο των θυρών, οπότε θα περιμένουμε 2-3 λεπτά και όσοι δεν ε, συμμετέχουν στην Κυκλισμένα των θυρών συνεδρίαση παρακαλούνται να εξέλθουν.